Friends, we start the meeting and hopefully all those... Αρχίζουμε αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω ότι ήδη έχουν έρθει αυτοί που πρέπει για τις ψηφορίες. Ελπίζω ότι έχετε καθίσει και έτσι μπορώ να ξέρω ποιος είναι πού. Να ξέρω δηλαδή ότι ο σωστός άνθρωπος βρίσκεται στο σωστό έδρανο και ψηφίζει. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε λάβει ένα μήνυμα από τον Τόμας Χέντελ και θέλω να σας ευχαριστήσω διότι τον υποστηρίξατε και θα παραμείνει πρόεδρος της Επιτροπής. Ακόμη δεν είναι θέση να έρθει στο Κοινοβούλιο. Τώρα πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία σε αυτή τη φάση. Αλλά έχει βάσει με ελπίδε ότι σε ένα-δύο μήνε θα βρίσκεται ξανά εδώ. Αυτό ήθελα να σα πω. Κάποιοι ε, από εμά τελευταίου μήνε είχαμε κάποια άμεση επαφή μαζί του. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελε να μας πει. You put them in the right place. Uh... Ελπίζουμε ότι έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Uh, uh, Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Έχουμε την γνωμοδότηση για την απαλλαγή 2015 του Γενικού Υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αρχίζουμε από την πρώτη συμβαστική. ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 4. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Έλεγχος για τη συμβαστική υπαριθμών φαίνεται. Ψηφίζω. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Θέλετε να το δείτε, το νούμερο. Να είναι γραμμένο. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για το 18. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Μπορούμε να ξαναδούμε το αποτέλεσμα. Α, πρέπει να γίνει η επανάληψη της ψηφορίας για το 18. Ψηφίζουμε. Is now ψηφορίας. 18. Απορρίπτεται. 26 ψήφι κατά. 21 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψήφισαμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Λείπουν για δύο ε, ψήφι, αλλά τόσο δεν πειράζει και εγκρίνεται 46-4. Χάρκιν. Ευρωπαϊκό Κέντρο για Ανάπτυξη Κατάρτιση ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Σχυρία Χάρκιν. Υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η πρώτη τροπολογία ήταν αυτή. Πρώτη τροπολογία επαναλαμβάνει. Ψηφίζουμε για τον έλεγχο. Πέρα ψηφοφορία. Και απορρίπτεται με 27-19. Πρώτη συμβαστική υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 είναι προφορική Μπασίρ και συγκεντρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 χωριστή ψηφορία. πρώτο τμήμα τονίζει ότι έγινε προσαρμογή των ιστών προς τα κάτω υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Διορθώνει πρόεδρος Χάρκιν 13. Υπέρ, κατά, απόχέ συγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Όπως τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους. Συγχαρητήρια κυρία Χάρκιν. Τώρα πάμε στην απαλλαγή για το Eurofound. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Δεύτερη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες μέχρι το 9. Ψηφιστεί μαζί με το 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...18 με 19 που εγκρίνεται 20 και 21 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και το σύνολο τώρα της γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 8 ψήφους. Επόμενη απαλλαγή. Χάρκιν. Για το EU όσα πρώτη τροπολογία μαζί με την υπερθμόν 2 για την Εμείς υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Τρία. προφορική τροπολογία της κυρίας Τόμτς και της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Ένα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 48-3. Απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ETF Harkin. Πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την πρώτη τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι καταπίπτει, διορθώνει ο πρόεδρος. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε το 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 με την 8 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 5 9, ε, συγγνώμη. εννέα μαζί με την... Όχι, εννέα μόνη τη διορθώνει η πρόεδρο. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτωτα. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα Τις γνωμοδότησης ψηφίζουμε πέρασε. Με 46 ψήφους εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την γνωμοδότηση για την ε, απαλλαγή που αφορά τους οργανισμούς της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015. Συμβαστική υπερθυμών 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη συμβιβαστική 3 ψηφίζουμε όσον αφορά την συμβιβαστική 3 πέρας εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ Προπολογίε 9 και 10 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Με 43 ψήφους εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότηση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. το έφυσε. Πρώτη συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 12. Ψηφίζουν. Πέρα τη ευφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 13. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος για το 13. Ψηφίζουμε. 13. Πέρασε. Shall we wait for her? Θέλετε να περιμένουμε. Αν βιαστείτε, θα κάνατε διαφορά ίσως. Αρχίζουμε από την αρχή. Τροπολογία 13. Πρέπει να πατήσετε άλλη μια φορά τα κουμπιά. Πέρας ψηφοφορίας. Έλα μου Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 103, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 41 ψήφους υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. σχέδιο γνωμοδότηση για τις διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και Τρίτων χωρών. Έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον της Χέλγκα Στίβενς και αρχίζουμε. Τροπολογία Δύο, 20 και 21 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 και 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 5 και 29, 30 και 31. Okay. We vote on amendment 30. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. Όχι. Θα πάμε στην 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω πως πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 8 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 31 ψήφους κατά. 9 υπέρ κατά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 Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 49 ψήφους υπέρ. Και καμία ψήφο κατά. We move on to um, uh, the uh, Helga Stevens report. Περνάμε στην έκθεση της Helga Stevens. Σχέδιο γνωμοδότηση για επιτρεπόμενε χρήσει έργων ή άλλων αντικειμένων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Αρχίζουμε με τη συμβιβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά τις αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Τροπολογίες 2, 16 και 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε. Υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, 26 και 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελευταία τροπολογία 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το συνολικό σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 49 ψήφους υπέρ. that all? Okay, that was the voting session. Τελείωσε η ώρα των ψηφοφοριών. Yeah.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 καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας, τροποποίηση της οδηγίας 2004 κάθετος 37, να αρχίσω λέγοντας κάποια εισαγωγικά. Ε, είμαι εισηγήτρια εδώ να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη σκληρή δουλειά τους και τις ε, επικοδομητικές τροπολογίες και τροποποίησεις. Είναι σίγουρα κάτι δύσκολο, το θέμα είναι πολύ τεχνικό και υπήρχαν πολλές εντελώς διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους στηρίξατε τις τροπολογίες μου Πολλοί από εσάς υπέβαλαν εκ νέου τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ε, όλους εσάς για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται επαρκώς από αυτές τις ουσίες. Και η οδηγία για τα χημικά δεν είναι ε, δεσμευτική ως προς τις ανώτατες τιμές και δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι, δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης. Ε, βέβαια δεν, ψάχ, δεν σκοπεύουμε να προστατεύσουμε μόνο τις εγκύους αλλά όλους τους εργαζόμενους. Ε, πάνω από 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολούνται σε τομείς που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία και υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα. Η Γαλλία και η Γερμανία, ας πούμε, έχουν θέσει ανώτατα ε, όρια στις τιμές αυτών των ε, ουσιών. Εάν καταφέρουμε τώρα να συμφωνήσουμε γι' αυτό το θέμα και για τις ρήτρες αναθεώρησης, θα καταφέρουμε να χτενίσουμε το κείμενο και να κάνουμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις ε, τεχνικού χαρακτήρα. Εδώ έχω και ένα άρθρο που αναφέρεται, ε, μάλλον ένα ρεπορτάζ για ένα εργοστάσιο παραγωγής λίκρα στις κάτω χώρες, όπου αυτή τη στιγμή έχει, ε, οι εργαζόμενοι έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με την Dupont για την εταιρεία παραγωγής, διότι έχουν γεννηθεί πολλά παιδιά από εργαζόμενες σε αυτό το εργοστάσιο, τα οποία έχουν σοβαρές αναπηρίες. Και υπάρχει άμεση σχέση των ε, προβλημάτων αυτών με τα χημικά στο εργοστάσιο. να πω πως θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες δικές σας στην έκθεση και να πω πως ε, αρκετές τροπολογίες είναι πολύ ισορροπημένες, λαμβάνουν υπόψη την ε, οπτική γωνία πολλών ενδιαφερόμενων φορέων και φυσικά αυτή η Επιτροπή είναι δεσμευμένη σε πολιτική που βασίζεται σε στοιχεία. Αυτές όμως οι ανώτατες τιμές δεν αφορούν μόνο τα ασφαλή όρια. Όπως ε, είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε 100% την ασφάλεια των εργαζομένων είναι να κλείσουν τελείως τα εργοστάσια τα οποία χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες. Αυτό βέβαια δεν είναι ρεαλιστικό και επειδή εμείς είμαστε πραγματιστές στην Επιτροπή προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι ε, μπορούμε. Αυτές οι ανώτατες τιμές είναι ε, μία μέση λύση ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι πολιτικό το θέμα επίσης και πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία. Φυσικά και θα ακούσουμε τις απόψεις όλων, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουν ε, υποφέρει, έχουν πληγεί από αρρώστιες, από καρκίνους που οφείλονται σε αυτές τις ε, χημικές μεταλλαξιακόνες ουσίες, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να ε, πληρώσουν ιατροφαρμακευτική αγωγή και τους οφείλουμε τη βοήθειά μας. Ε, οφείλουμε επίσης να σταθούμε δίπλα σε όλους ε, τους ασθενείς, όλους ε, όσοι νόσησαν εξαιτίας της δουλειάς τους. Και αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλους. Είναι εν τέλει μια πολιτική απόφαση. Και θα ήθελα τέλος να πω πριν δώσω το λόγο στους ότι υπάρχει και ε, μία νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει ένα σύνολο πρόσθετων χημικών ουσιών. Και να πω πως με εξέπληξε αυτό, διότι όπως έχουμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή, αυτό αυτή η νέα δέσμη, των νέων σύνολο ουσιών δεν είναι τόσο φιλόδοξο όσο μας είχαν υποσχεθεί και όσο περιμέναμε. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε διαβεβαιώσει ότι η νέα ομάδα ουσιών θα καλύπτει τις διπλάσιες ουσίες από ό,τι η προηγούμενη. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει ακολουθώντας αυτή τη φιλόδοξη πορεία της για να συμπεριλάβει έτσι όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις ουσίες. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και θα αρχίσω από τον κύριο Ρολάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντως είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Θέμα σημαντικό για τους ε, έμιστους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να, να ζητήσουν λύση και συνένεση για το ζήτημα αυτό. Και θα πρέπει έτσι επομένω η πολιτική προστασία τη υγεία των εργαζομένων. Θα πρέπει να προ αυτή την κατεύθυνση. Αν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια συνένεση, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη και δύσκολη να επιτευχθεί ισορροπία. Και εγώ έχω ήδη υποβάλει κάποιε τροπολογίε και έλαβα υπόψη την Επιστημονική Επιτροπή αλλά και την Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα υγεία. Και ε, ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Εκεί συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και τα κρατημέλη. Οπότε κάθε φορά ε, αν κάποια λύση, δεν συμφωνούν βέβαια για όλα. Διαφωνούν επίσης ε, οι επιστήμονες μεταξύ τους, όπως διαφωνούν και οι κοινωνικοί εταίροι για ορισμένα θέματα. Άρα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις προτάσεις μας, παρά το ότι εκείνοι δεν τα έχουν βρει. Δεν θα σας λέω μία-μία τι τροπολογίε εγώ. θα πρέπει πάρα πολύ χρόνο. Για αυτές τις τοξικές ουσίες είπαμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και για τη σκόνη ξύλου. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει λόγος διάκρισης μεταξύ αυτής της σκόνης όταν είναι μαλακό το ξύλο ή όταν ε, υπάρχουν άλλου είδους ε, υφή του ξύλου. Πάντως δεν συμφωνούν, είπαμε οι επιστήμονες. Εγώ θα συμφωνήσω με τους κοινωνικού εταίρους. 3 μιλιγκράμμ ανακυβικό, λέγονται σαν οριακή τιμή. Και θα πρέπει μετά από 5 χρόνια να γίνει αναθεώρηση, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς να πλησιάσει την ε, οριακή τιμή που θέλουν οι επιστήμονες. Όλα αυτά εξελίσσονται γιατί έχουμε συνέχεια καινούργια μόρια, έχουμε καινούργια προϊόντα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, άρα πρέπει να παρακολουθούμε. Το κόμμα 6 είναι θέμα εδώ του Συμβουλίου, είναι περίπου 10 χώρες που έχουν τοποθετηθεί και συμφωνώ με τη γνώμη αυτήν. κρυσταλλική ουσία τέλο πάντων θα πρέπει να συμφωνήσουμε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ε, αυτοί που ασχολούνται με το θέμα κάποιοι στην πράξη θα πρέπει να τους ακούμε. Άρα αυτό θα κάνουμε για αυτό το 1 μιλιγράμμα ένα κυβικό μέτρο. Πρόκειται κάποια προληπτικά μέτρα ε, που είναι συνοδευτικά και καθώς επίσης έχουμε και την ε, καλή πρακτική για να μην υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες για τους εργαζόμενους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εξουσιοδότηση πράξης αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αυτό γίνεται συνήθως για πράγματα που δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά ενώ τώρα αντιθέτως έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα. Συμφωνώ με την πρόεδρο μας. Περιμέναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει περισσότερες προτάσεις. Ε, δεν ξέρω θα είναι το δεύτερο ε, γύρο, αλλά για τον πρώτο γύρο ξέρουμε. Είναι υψηλά ο πύχης των προσδοκιών. Να δούμε τι θα κάνει στο μέλλον η Κομισιόν. Πάντως, Εγώ είμαι στη διάθεση όποιου θέλει να τα συζητήσουμε, μια που τα θέματα είναι περίπλοκα. Δεν μπορούμε να τα πλουστεύσουμε. Και ελπίζω ότι και η Πρόεδρος και οι άλλοι σκιώδες ηγητές θα μπορέσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να καλύψουμε τις ανησυχίες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ε, Επίση, ελπίζω ότι τελικά θα συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ μια δεκαετία που δεν έχει σημειωθεί πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μάκιντάιρ είναι ισχυρή για το ECR, δεν είναι όμω που σιάζει. Κυρία Χαρτ, μήπω θέλετε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος κυρία Μακιντάρη θέλει να ζητήσει συγγνώμη για την απουσία της και μου ζήτησε να παρουσιάσω την ε, δική της άποψη. Έχουμε, προτείν, έχουμε λάβει προτάσεις για διαφορετικά ανώτατα όρια, διαφορετικές ανώτατες τιμές και αυτή την πρόταση την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Όμως αυτές οι ενότητες τιμές πρέπει να είναι αναλογικές και να έχουν προκύψει μετά από επιστημονική ανάλυση. Η κυρία Μακιντάρη λοιπόν είναι της άποψης ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποφύγουμε να προτείνουμε όρια τα οποία είναι ανέφικτα. Για παράδειγμα, κρυσταλλικό πυρίτιο, διοξίδιο κρυσταλλικού πυριτίου. Εδώ το ε, όριο που έχει προταθεί είναι 0,005. Δεν είναι εφικτό. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος μέτρησης που να μπορεί να μετρήσει μετρήσει τόσο χαμηλή τιμή. Δεν είναι λοιπόν ρεαλιστική αυτή η πρόταση. Έπειτα, ορισμένες χημικές ουσίες οι οποίες είναι τοξικές για, την, ε, για το αναπαραγωγικό σύστημα. Η έκθεση σε αυτές τις ουσίες πρέπει φυσικά να συρρυκνωθεί, να μειωθεί και αυτό ε, θα γίνει μέσω της μείωσης του χρόνου έκθεσης της ουσίες αυτές. Μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε μείωση των ανώτατων τιμών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πιέσουμε την Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε όμως εδώ να προτείνουμε ανώτατα όρια τα οποία είναι τόσο χαμηλά που δεν είναι πλέον ρεαλιστικά. Ήδη υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές οι οποίες προστατεύουν τους εργαζόμενους. Το ζητούμενο πιστεύω εδώ θα έπρεπε να είναι να ε, μειωθεί ο χρόνος έκθεσης στις ουσίες αυτές και πρέπει να ισχύει αυτό για όλους τους εργαζόμενους. Όμως για να γίνει ε, αυτό το βήμα πρέπει πρώτα να ε, γίνουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε όλους τους εργαζόμενους. Ούτε αυτό είναι ρεαλιστικό διότι θα επιβαρυνθεί υπερβολικά ε, το σύστημα υγείας στην κάθε χώρα. Και χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική λύση. Μία θα μπορούσε να είναι η πρόληψη και υπάρχει μια τέτοια αναφορά σε μια αιτιολογική σκέψη, αλλά και πάλι δεν ξέρω πώς μπορούμε ρεαλιστικά να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση. Μετά, οι μετρήσεις. Και ο καθορισμός τόσο χαμηλών ανώτατων ορίων καθώς και τόσο χαμηλού χρόνου έκθεσης πιστεύω πως είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που είναι ανέφικτο να εφαρμοστούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ. Κυρία Βέπερ, έχετε το λόγο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι έχει τεράστια σημασία το θέμα που συζητούμε. Και το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Πολύ περισσότερο από το να αναζητούμε μετά εξειδικευμένη βοήθεια θεραπεία. Και υπό αυτό το πρίσμα εγώ αναζητώ ποιος είναι ο βελτιωστός τρόπος να νομοθετήσουμε. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πολύ καιρός για να μην έχουμε αναθεωρήσει κάτι τόσο σημαντικό, δεδομένης μάλιστα της ταχύτητας της επιστημονικής πρόοδου. Ταυτόχρονα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει τρία διαφορετικά πακέτα. Συμφωνούμε, καταλαβαίνουμε γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε στα χέρια μας επιστημονικές μελέτες αλλά επίσης πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη, στην πραγματικότητα. Έχουν ε, διενεργηθεί πολλές επιστημονικές μελέτες και μάλιστα χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο του ευνομοθετήν λοιπόν δεν θα έπρεπε να φροντίζουμε να μην ξοδεύουμε χρήματα δυο φορές, τρεις φορές για την ίδια αξιολόγηση. Με αυτά ως δεδομένα εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία ε, συνένεση στο Κοινοβουλίο μας να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ε, του κανονισμού με αυτή την αναθεώρηση του. Εάν ε, κανείς κοιτάξει στις τροπολογίες, πολλές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την... μάλλον έχουν σχέση, ακολουθούν την κατάσταση που ισχύει σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη στη χώρα του προτείνοντος, γιατί τα όρια είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα και πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να συμφωνήσουμε. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει η συμφωνία να συμπεριλάβουμε ορισμένες τοξίνες, αλλά ε, πρόκειται για ουσίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις καρκινογόνες. It's important to have them uh, there. Um... Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι η εφαρμογή αυτής, αυτού του κανονισμού, αυτών των πρότυπων. αυτής της μάλλον. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τα όρια στο χαρτί, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται στην πράξη. Νομίζω θα τα συζητήσουμε αυτό το θέμα ζήτημα τη εφαρμογή πιο αναλυτικά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τι τροπολογίες. Υπάρχει ένα θέμα όπου εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα, τι θα γίνεται. Και αυτό είναι η διαρκής παρακολούθηση του, της υγείας του εργαζόμενου. Και μάλιστα ακόμα και όταν φύγουν από τον χώρο εργασίας. Γιατί φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο, είναι πολύ πιθανό μάλιστα, η επιδείνωση της υγείας να έρθει πολύ αργότερα, πιο, πιο μετά από την ε, αποχώρηση του εργαζομένου. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους εργοδότες, από τις εταιρείε να κάνουν αυτή την παρακολούθηση ή μήπως τελικά αυτό είναι μέρος του, ε, του ε, συστήματος υγείας μιας χώρας, του κρατικού συστήματος υγείας, δηλαδή το κράτος να έχει τους μηχανισμούς για να ελέγχει την υγεία των πολιτών του, για να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας των εργαζομένων σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτά τα πράγματα Ελπίζω να τα διευκρινίσουμε στις συζητήσεις μας όταν συναντηθούμε για τα, τις τροπολογίες. Χρειάζεται να τα γνωρίζω αυτά γιατί ε, διαφορετικά πώς θα ε, συγκεντρώσω εγώ και την υποστήριξη της ίδιας της πολιτικής μου ομάδας. Πρέπει να ξέρω τι θα τους πω, τι θα τους ζητήσω. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα θέμα στο οποίο οφείλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, να πάμε μπροστά. Thank you. Uh, is uh, Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ. Ο σκιώδης συζητητής δεν είναι εδώ. Επομένως θα δώσω το λόγο στους πράσινους. Καρίμα, Καρίμ Ατέλ. Επουσιάζει και αυτή. Η κυρία Άκα. δεν είναι εύκολο κανείς να δουλέψει και να πιάσει τόπο η δουλειά του για την αναθεώρηση αυτού του νομοθετήματος γιατί η στόχη για τα καρκινογόνα ήταν η εξή. Να μπορέσουμε να καλύψουμε πρώτα πρώτα τι γίνεται με τη σκόνη από τους κρυστάλλους του πυρητήρου. Να μπορέσουμε να καθορίσουμε μια οριακή τιμή σε σχέση με την τρίτη ενότητα. Ή στο τρίτο παράρτημα τέλος πάντων. Εδώ υπάρχουν πολλές δυσκολίες που συναντά κανείς σε αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάποιο είδους μεθοδολογία που να μπορεί να πιάσει τόπο. Να σας εξηγήσω τι εννοώ δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον κύκλο παραγωγής όσον αφορά την σκόνη από αυτούς τους κρυστάλλους. Δεν ξέρουμε να υπολογίσουμε τι απόσταση κάνουν αυτές οι ουσίες, αυτές οι σκόνες. και αν ε, έπρεπε να προχωρήσουμε στο να δούμε πώς θα περιούσουμε αυτή τη σκόνη που είναι το λογικό, αυτό θα ήταν μεγάλη δαπάνη. Γιατί στα εργαστήρια ποτέ δεν το σκέφτονται αυτό, να κάνουν δηλαδή κάποιο είδους επενδύσεις για μια τέτοια προσπάθειες για να υπάρξουν και κάποια κίνητρα από το κράτος. Ενώ θα είχε αυτό αποτελέσματα. Προσπάθησα να βρω λοιπόν μια άλλη λύση που να ε, είναι πιο βιώσιμη. Να δούμε πώς θα υπάρχει η ατομική προστασία. Γιατί η συλλογική προστασία κατά κάποιο τρόπο για την εταιρεία είναι κάτι που δεν είναι βιώσιμο πλευράς δαπανών. Δεν δίνονται κίνητρα. Και εντωμεταξύ να προχωρήσουμε προς την ε, απαγόρευση των ε, τοξικών αυτών των ουσιών τέλος πάντων και ταυτόχρονα να έχουμε προστασία ατομική των εργαζομένων. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι αν εντόπισαν ε, κάτι για την ατομική προστασία στο κείμενο της οδηγίας, εγώ δεν το βρήκα και να μην ξεχνούμε ότι όταν έχουμε τους θανάτους από τον αμύαντο, πολλές φορές έχουμε και τη, τους συζύγους των εργαζομένων. Γιατί, γιατί τους είχαν πλύνει τα ρούχα Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια λύση ε, βιώσιμη, θα, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση μέχρι ότου η οδηγία καταλήξει σε κάποιες οριακές τιμές. Τα ε, σώσαμε έτσι ζωές. Λέμε τώρα τι ισχύει για αυτές τις οριακές τιμές, για ε, τη σκόνη από σκληρό ξύλο και έλεγε αυτή η πρόταση ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακέ τιμέ στα βρετματρία. Γι' αυτό το χλωριούχο βινίλιο και από τη σκόνη του σκληρού ξύλου στο σχετικό παράρτημα. Και έχουμε από την Επιτροπή Σκόλα για το 2002-2004, αυτή η Επιτροπή τέλο πάντων έλεγε ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι οριακέ τιμέ. Άλλο θέμα τη οδηγία να καθορίσει τις ουριακές τιμές για 10 καρκινογόνες επιπλέον ουσίες. Όμως δεν προχώρησε αυτή η φιλοδοξία, αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη. Δεν είναι δέκα αυτές οι ουσίες, είναι πολύ περισσότερες. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Άλλες δύο αναθεώσεις θα πρέπει να γίνουν για να προσθέσουμε και άλλες καρκινογόνες ουσίες. Σαν να λέμε στους εργαζόμενους, δηλητηριαστείτε εσείς όσο εμείς ψάχνουμε. Ε, όχι, πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένε, βιώσιμες και υλοποιήσιμες. Θα πρέπει βέβαια και οι επιχειρήσεις με όλες αυτές τις προσπάθειες να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το στρίμωγμα που υπάρχει. Και ακριβώς επειδή είναι τέτοια η συγκυρία, οι επιχειρήσεις κάνουν περικοπές στα θέματα ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Πάντοτε είναι θέμα σημαντικό, πάντως η σωστή ενημέρωση. Οι επιδημιολογικές μελέτες για να καταλάβει κανείς τι γίνεται εκεί στο χώρο εργασίας. Όμως δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες. Να, για τον αμύαντο ξέρουμε τι έγινε τόσα χρόνια. Δεν έγινε έρευνα εις βάθος για τη θεραπεία. ε, λαμβανόταν υπόψη μόνο συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, αρρώστιας των και όχι πολλές άλλες δεν τις απέιδαν τις, τα, τα, άλλα, τα άλλα συμπτώματα στον αμύαντο. Αλλιώς θα ε, μελετούσαμε όλα τα σενάρια. έχουμε ας πούμε τώρα καταλήξει ότι υπάρχει αρρώστια που έρχεται από τους κρυστάλλους του πυρητίου, αλλά έχουμε και άλλες πολλές ασθένειες. Άρα χρειάζεται έρευνα και θα πρέπει να γίνει η μετάβαση προς έναν καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος βιώσιμο και αποτελεσματικό. Εγώ να την Κομισιόν πιο άρτιο έργο και όχι τόσο αποσπασματικό, εμβαλωματικό. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Αν κάποιος εκτεθεί σε καρδιογόνες ουσίες, ε, βέβαια μακροπρόθεσμα πρόκειται να έχει πρόβλημα υγείας. Και υπάρχουν οι μέθοδοι. Προχωρούμε προς την κατάργηση αυτών των ε, ουσιών. Αλλά εκτός από αυτά τα υλικά που έχουμε επισημάνει υπάρχουν και άλλα όπως υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των βλαπτικών και δεν επιφέρουν ε, προβλήματα στην υγεία του εργαζομένου. Merci, Κύριε Μέλα, σας ευχαριστώ. Στο θέμα αυτό έχουμε πάρει πολλές, πολλές εξελίξεις, αλλά και πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινίσουμε. Πρώτον, ποιος είναι ο στόχος του έργου μας. Μας ε, ζητείτε η γνώμη μας για μέτρα ε, που είναι προτεραιότητα που και πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες μάλλον για αυτά τα μέτρα. Η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να βρούμε ε, ουσίες και υλικά για να αντικαταστήσουμε αυτές τις ουσίες τα καρκινογόνα υλικά. Αυτό είναι το πρώτο. Η δεύτερη προτεραιότητα, εάν αποδειχθεί ότι είναι αδύνατο να αντικατασταθούν κάποιε ουσίε υλικά, είναι να, θέσουμε, να βρούμε τρόπου προστασία των εργαζομένων. Και σε τρίτη προτεραιότητα, να συζητάμε για το ζήτημα τη δοσολογία τη επιτρεπτή. Γιατί και αυτό. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πρόκειται τέ για ασθένειες που προκαλούνται από αυτές τις ουσίες, οι οποίες ε, ε, συνδέονται με πολλούς παράγοντες, είναι πολύ παραγωγικέ. Ε, αυτό ισχύει για όλα τα, τους καρκίνους, για όλα τα νεοπλάσματα. Επομένως, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ποιος παράγοντας προκάλεσε τι. Ε, αναφερόμαστε στην συμπερίληψη των τοξικό, ναι, των τοξινών που επηρεάζονται από την αναπαραγωγή και τη συμπερίληψή τους στους καταλόγους αυτούς. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες από αυτές τις ουσίες συνδέονται με καρκίνο ή με προβλήματα στην αναπαραγωγική υγεία, χωρίς να είναι πάντοτε όμως ξεκάθαρο ε, μάλλον είναι πάντοτε ξεκάθαρο αυτή τη ουσία προκαλούν προβλήματα στον απαραγωγικό σύστημα χωρί να ξεκάθαρο μετά από ποια δόση ε, οδηγούμαστε σε καρκίνου και μεταλλάξει. Εδώ χρειάζεται να ακολουθούμε τις επιστημονικές μελέτες ε, ε και η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι αυτό που χρειάζεται να ακολουθούμε είναι η αρχή της προφύλαξης και αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ουσίες οι οποίες δεν αναφέρονται στην έκθεση ε, και έχουν ακουστεί 6-7 οι οποίες θεωρούνται καρκινογόνες σε ορισμένα κράτη-μέλη και όχι σε όλα θα θέλαμε αυτές να καλύπτονται σε μελλοντικές εκθέσεις. Επομένω, αυτή ο κατάλογο των νησιών θα πρέπει να ε, πηγαίνει πάντα προ τη διεύρυνση. Τίθενται μια σειρά προβλημάτων που έχουν σχέση με τα μέτρα που ζητάμε. Γιατί τα μέτρα που ακολουθούνται δεν είναι ίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις το όριο είναι που ζητείτε είναι υπερβολικά χαμηλό. Και αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα για ουσίε οι οποίε ε, μάλλον, τα οποία συνδέονται με πολλέ θέσει εργασία. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας, ε, ε, η σκόνη του ξύλου, για παράδειγμα, όταν έχουμε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε χρησιμοποιούν και γνωρίζουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα πρότυπα τα δικά τους δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα δικά μας. Και γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες εργασίας στις χώρες αυτές είναι απαράδεκτες και από ιατρικής και από νομικής απόψεως. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ελπίζω λοιπόν έχοντας κάνει αυτές τις μικρές παρατηρήσεις ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία στη συζήτηση αυτή. Ε, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικός ο ρόλος μας. Ε, θα ε, έπρεπε, με, με, εκπλήσει μάλλον το γεγονός ότι έχουμε περάσει μετά ε, τόσο καιρό προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μια μεγάλη έκθεση για όλες τις ενδιαφέρουσες, για όλες τις σημαντικές ε, ουσίες, ενώ θα ήταν ίσως καλύτερα να είχαμε πολλές μικρότερες θέσεις κάθε 6 μήνες, πιο τακτικά προχωρώντας. Ε, με αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να πω ότι θα προσβλέπω στη συνεργασία με τους ε, συγγενείς Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπαχ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την απόψή μου πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Πολλά από τις προτάσεις είναι αρκετά ε, φιλόδοξες, αρκετά γενναίες, όμως η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε ούτε τι μας περιμένει, ούτε πότε μας περιμένει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα εδώ. Τώρα, επιπροσθέτω, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο είναι ακόμα πιο επιφυλακτικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε, εδώ μεταξύ, την θέση τους και την άποψή τους και ακριβώς για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι εμείς ως ε, Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή, ως ε, Πρόεδρος εσείς κύριε Πρόεδρε και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ γενναίοι, πάρα πολύ φιλόδοξοι για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη από τα άλλα θεσμικά όργανα. Και να πω ότι αυτό το θέμα μου θυμίζει πολύ το σκάνδαλο με το ντίζελ. Γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα, γνωρίζουμε ποιες είναι οι βλαβαρές επιπτώσεις, έχουμε συζητήσει για ανώτατες τιμές, για χρονικό χρονοδιάγραμμα και χρονό έκθεσης και όμως ε, πρέπει να ε, καταλάβουμε επιτέλους ότι όσο καιρό συζητάμε αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, ασθενείς, έχουν νοσήσει από αυτές τις ουσίες και πρέπει πιστεύω να επικεντρωθούμε στο πραγματικό σκάνδαλο γιατί αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Τώρα, Νομίζω πως ε, στα επιμέρους θέματα για την τοξικότητα στην αναπαραγωγική υγεία είμαστε εντάξει. Θα μπορούσαμε βέβαια να δούμε το θέμα ίσως λίγο πιο επιστημονικά ή από την άλλη πιο συναισθηματικά. Όμως ε, θεωρώ πως πρέπει να ακολουθήσουμε την παρούσα οδό. Να βασιστούμε δηλαδή σε επιστημονικές μελέτες, σε ε, επίσημα στατιστικά στοιχεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και να χρησιμοποιήσουμε κάποια παραδείγματα των τιμών που έχουν ήδη τεθεί και να αναγνωρίσουμε ε, ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία έχουν, πολύ, ε, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχουν θέσει πολύ καλά πρότυπα ε, και παρά να αναλωνόμαστε στο τι είναι ρεαλιστικό, εφικτό και τι όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλη αυτή η συζήτηση νομίζω πως μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Θέλουμε όλοι το καλύτερο δυνατό, να ε, οδηγηθούμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Βέβαια, η εισηγήτρια με την τροπολογία 21 για τις ανώτατες τιμές κεραμικών ε, ινών νομίζω πως προτείνει μία περαιτέρω μείωση μίας τιμής η οποία όμως έχει ακριβώς τις ίδιες επιπτώσεις ε, σε σχέση ε, με άλλες ουσίες που έχουν μεγαλύτερο κόστος. Τα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να είναι κάπως ε, κοινικά, αλλά σε αυτά διαβάζουμε πως ο αριθμός των θανάτων από αυτή την ουσία είναι μηδέν. Και ε, βλέπουμε όμως παρόμοια τιμές και για άλλες ουσίες. Ε, αυτό που πρέπει να δούμε είναι και το κόστος για τους ε, εργοδότες και το κόστος για τους εργαζόμενους. Για τους εργοδότες μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετο κόστος αν αλλάξουν οι τιμές. Και νομίζω πως εάν ε, δεν αλλάξουν οι επιπτώσεις ε, στην υγεία με το να μειωθούν περισσότερο τα ανάτατα όρια, νομίζω πως δεν πρέπει να επιφορτήσουμε με ακόμα περισσότερο κόστος ε, την ε, βιομηχανία. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω, να παρακαλέσω μάλλον την εισηγήτρια να επανεξετάσει το θέμα για την τροπολογία 21 και ε, να επαναξετάσουμε την κατηγορία 1, 2, 3 όπου παρατηρούνται ακριβώς οι ίδιες επιπτώσεις στην υγεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, μια και δεν βρισκόμαστε ακόμα σε τελικό στάδιο, δεν έχουμε αποφασίσει ποια μορφή θα έχει το έγγραφο που θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι έχουμε προτείνει, ανώτατα όρια, ουσίες κτλ. είναι πράγματα τα οποία σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ήδη δρομολογηθεί, ήδη εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, για να βγούμε και παραέξω; Υπάρχουν, υπάρχει σχετική νομοθεσία. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά δεν διαλέξαμε στην τύχη κάποιες ουσίες, δεν τις βγάλαμε από το μυαλό μας. Και πρέπει να προσέξουμε στη σύγκριση με άλλες ε, χώρες στον κόσμο να μην βρεθούμε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε να προστατεύσουμε την υγεία. και σίγουρα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Δεν νομίζω πως εδώ υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων, κάποια αντίθεση στις απόψεις των μελών μας. Δεν ξέρω αν συναγωνιζόμαστε, ανταγωνιζόμαστε άλλες χώρες ή αν θέλουμε να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, πάντως ε, δεν θα έπρεπε να πασχίζουμε να φτάσουμε στον πάτο. Καλύτερα να στοχεύουμε προς την κορυφή ή έστω στη μέση σε τη φορά που κάνουμε. Και νομίζω όπως άκουσα πιο πριν, θα ήθελα και εγώ να μάθω γιατί υπάρχουν κάποιες προσθήκες, κάποια έξτρα παραπάνω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα και εγώ να μάθω τι θα γίνει με τις επόμενες ομάδες ουσιών. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε λίγο για να μας πει τι σκοπεύουν να κάνουν και να μας ε, δώσουν τη δική τους άποψη για το πώς μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές και ταυτόχρονα φιλόδοξοι να ενημερώσω επίση πω τι ερχόμενε εβδομάδε θα γίνουν κάποιε συναντήσει των σκιωδών εισηγητών. όπου θα προσπαθήσουμε και να είμαστε ρεαλιστές, αλλά και να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη θέση. Διότι δεν μπορεί η Ευρώπη να βρίσκεται στο τέλος, στην τελευταία θέση του καταλόγου. Αυτό φανταστείτε τι επιπτώσεις έχει και στην αγορά εργασίας και στο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πεθαίνουν από καρκίνους που οφείλονται στο χώρο εργασίας τους. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μας συζήτηση για αυτό το θέμα. Νομίζω πως έχουμε όλοι την ίδια ή παρόμοια άποψη. Θέλουμε το ίδιο. Είναι σίγουρα θέμα υψής της προτεραιότητας η υγεία στο χώρο εργασίας. Και αν μου επιτρέπετε, θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα και να δούμε και το πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Παρακαλώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Σιγητρία. κυρία Σιγητά. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για το πολύ καλή δουλειά που έχετε προετοιμάσει, την θέλησή σας να προχωρήσει η συζήτηση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μας καθησυχάζει. Το χαιρόμαστε για το γεγονό ότι συμφωνούμε σε ότι χρειαζόμαστε ένα φιλόδεξο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Πρώτον, να σχολιάσω κάτι που συζητούσατε πριν Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί γρήγορα η συζήτηση για αυτό το πρώτο πακέτο. Γιατί όπως είπατε πράγματι αυτή η συζήτηση είχε καθυστερήσει, αλλά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Ζητείτε από την Επιτροπή Μότου που υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα να ενημερώσετε τα σχετικά όρια και να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Όμως με το που συμβαίνει αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και την διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αμέσως μετά να κάνουμε και την αξιολόγηση αντικτύπου. Όλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρο. Και αυτό οδήγησε σε αυτό που επισημάνατε στις καθυστερήσεις, παρόλο που τώρα κινούμε γρήγορα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σύντομο να καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτό το πακέτο τώρα και παραμένει υποχρέωση τη επιτροπή να επαναξιολογεί τον κατάλογο και τα όρια με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά εξάλλου. Αξιολογούμε νέε ουσίες ή υλικά. Αναφερθήκατε στο δεύτερο πακέτο και στο γεγονό ότι αυτό το δεύτερο πακέτο ε, δεν συμπεριλαμβάνει όλε τι χημικέ ουσίε που θα περιμένατε. Πράγματι. Ο λόγο είναι ο ακόμα μια φορά. Χρειαζόμαστε να έχουμε ε, στέρεα επιστημονικά δεδομένα που θα να έχουν συζητηθεί στην τριμερή επιτροπή διαλόγου και να έχει ολοκληρωθεί και αξιολόγηση ενδεικτύπου. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δυστυχώς δεν είχε ολοκληρωθεί ε, για όλες, τις, για όλες αυτές τις ουσίες μέχρι τον Ιανουάριο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα νομικού ορισμού, νομικά προβλήματα ορισμού των χημικών νοσιών. Πάντως πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πιο αναλυτική παρουσίαση της πρότασης αργότερα. Πάντως, ε, να επισημάνω ότι έχει ε, ανακοινωθεί και, ε, ε, έχει δημοσιευθεί και ανακοίνωση της Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια, την ίδια ημερομηνία με το πρώτο πακέτο, τον Ιανουάριο δηλαδή, όπου και αυτή είναι, περιγράφει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος με ένα τρίτο πακέτο χημικών ουσιών στις αρχές του 2018, που ο κατάλογος τότε εκεί θα συμπεριλαμβάνει και νέες ουσίες, και νέες χημικές και ε, συμπεριλαμβανομένων και χημικών ουσιών που δεν είναι αναγκαστικά ή γνωστό αναγκαστικά ότι είναι καρκινογόνες, αλλά παρόλα αυτά για αυτές θα προταθούν ε, ενδεικτικά ανώτατα όρια. Ε, ακολουθείται η διαδικασία της επιτροπολογίας και αναμένουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτή τους επόμενους μήνες. Επόμενο μήνα. Και όταν είμαστε έτοιμοι αργότερα κάποια στιγμή ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας πιο αναλυτικά αυτό το δεύτερο πακέτο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζουμε, ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει. Άρα, εναγωνίως, περιμένουμε. συζητήσαμε, ακούσαμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε ρεαλιστές, αλλά έχουμε και φιλοδοξίες, γιατί πάρα πολλοί είναι Ευρωπαίοι που πεθαίνουν για αυτό το λόγο. Διότι έχουν εκτεθεί Χημικές ουσίες ή σε σκόνη. Και παθαίνουν καρκίνο. Και όλα αυτά στο χώρο εργασία. Και αυτό υπάρχουν διαφορέ μεταξύ κρατών μελών γιατί αλλού υπάρχει χαμηλό, αλλού υψηλό επίπεδο προστασία those uh, uh, regulations that we want to be the same for all of Europe. Uh, θα θέλαμε να υπάρχει ίδια ρύθμιση για όλη την ε, Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο σε κάποιες χώρες. Επιτρέπονται δηλαδή αυτά που κάνουν σε μερικές χώρες και μην επιτρέπονται αλλού. Γιατί είναι πιο αυστηρή νομοθεσία. Of, of support and regulation, of course. Uh, and we also know that uh, if we compare with what's in reach, if we compare... Σκεφτούμε τι λέει το reach, τι προβλέπετε στην Αμερικανική νομοθεσία. Βλέπουμε ότι εκεί είναι πιο ψηλό το επίπεδο προστασίας. To, um, uh, work. Περιμένουμε να συνιστή συνεργασία μα για το θέμα να υπάρξει ευρύτερη δυνατή συνένεση στην Επιτροπή μας. Και έτσι να πετύχουμε το στόχο μας. Θα είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνηθούμε και με τους σκιώδεις ηγητές και θα συζητήσουμε. Θέλει άλλο το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Εδώ δεν έχουμε και πολλές χημικές ουσίες. Κυρία Λαουρίστη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δε... Συνάδελφε, έχουμε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά κάποιο τρόπο αυτό όμως είναι λίγο μπαγιάτικο, γιατί αυτό το, έργο, το έγγραφο φαίνεται ημερομηνία Απρίλιο του 2016. Είστε Λίμπη, αλλά τώρα ε, βλέπουμε 15 σελίδες, από τις οποίες μόνο μια μισή ασχολείται με τους ανθρώπινους πόρους. 13,5 σελίδες ε, μιλούν για μηχανήματα, για τεχνολογία, δεδομένα κλπ. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή μας να βοηθήσει σημαντικά σε αυτή την έκθεση της Ήτρα με την γνωμοδότησή μας. Μεγάλη μου χαρά, εγώ ανέλαβα να συντάξω αυτή την ε, γνωμοδότηση. Γιατί πιστεύω στην ε, ψηφιοποίηση. Να δούμε αυτή τη μια μισή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαπιστώσουμε ότι ως επιτοπλίστων ε, σχολιάζεται η παιδεία, η ανάγκη για ε, εργαζόμενους με δεξιότητες, αλλά τίποτα δεν αναφέρεται για κοινωνική προστασία, τίποτα για όλα αυτά τα θέματα τα οποία στην Επιτροπή μας συζητούμε και τα θεωρούμε και τόσο σημαντικά. Τόνισαμε σε αυτά τα θέματα, θα τονίσουμε τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στην επασχόληση, τι πρέπει να κάνουμε στοχευμένα, στις σχετικές πολιτικές για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές μεταξύ χωρών και μεταξύ περιφερειών. Και όλα αυτά προς οφείλος των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών και των καταναλωτών που όλοι αυτοί συμμετέχουν στην ε, ψηφιακή οικονομία επίσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προβληματική για τις επιπτώσεις τη ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας, στην ε, δομή των διαφόρων επαγγελμάτων και τα προγνωστικά είναι καθόλου ρόδινα. Μιλάμε για 40-50% των επαγγελμάτων που θα εξαφανιστούν. Έτσι λέει ο, ο ΣΑ, ή τα λέει λίγο καλύτερα ο ΣΑ, αλλά υπάρχουν ε, διάφορες παραλλαγές λένε ας πούμε ότι θα αλλάξει η δουλειά, το καθήκον του εργαζόμενου, θα αλλάξει το περιεχόμενο του επαγγέλματο. Άρα θα πρέπει κανείς να αποκτήσει νέε δεξιότητες. Για να δούμε μόνο ποιοι θα πρέπει να καλυφθούν από αυτές τις αλλαγές. Κυρίως αυτοί που δεν έχουν υψηλέ δεξιότητες θα πρέπει να επανακαταρτιστούν και αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, κάτι άλλο που να πούμε στην γνωμοδότηση είναι η κοινωνική πρόνοια και προστασία. Αυτά που συζητούσαμε σήμερα το πρωί. Το πόσο αλλάζει η απασχόληση τι γίνεται με την ευάλωτη απασχόληση, τις νέες μορφές απασχόλησης, την απασχόληση με τις πλατφόρμες. Το και ακόμα δεν έχουν βρεθεί αυτές οι λύσεις και δεν προχωράει ο κοινωνικό διάλογος. Άρα εμείς εδώ θα κάνουμε τις προτάσεις μας σαν Επιτροπή. Να πούμε ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Επίσης υπάρχει πρόβλημα και με τα κοινωνικά δικαιώματα, για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ των εργαζομένων επιμέρους κλάδων σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί για κοιτάξτε τι γίνεται με τη νέα γενιά. Αυτοί έχουν πιο πολλές ψηφιακές δεξιότητες που αποκτούν στο σχολείο και τις σχολές όμως ε, έχουν κινητικότητα αλλά δεν μένουν εδώ, φεύγουν, πάνε στη ΣΥΠΑ, πάνε στην Κίνα α, μπορεί και να γυρίσουν αλλά δεν διανοούνται ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όταν γεράσουν με την υγεία τους κλπ. κλπ. Άρα και αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε. Η κοινωνική προϊόν για αυτούς, για αυτούς που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Είναι όμως δικό μας καθήκον. Επίσης, υπάρχει θέμα με τις δεξιότητες, με την κατάρτιση, γιατί πάρα πολύ συχνά υπάρχει το πρόβλημα των ψηφιακών δεξιότητων. Πολλές φορές το αυτό το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ τεχνοκρατικά, όπως και με την πληροφορική. Όμως ε, κάτι, κάτι, κάπως αγγίζει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα μεγάλα τα δεδομένα, τα μαζικά δεδομένα, big data. που σχετίζονται με πολλά μέρους προβλήματα για διαχείριση, για πολλά είδη επιχειρήσεων. Οπότε αυτό θα σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους θα πρέπει να προετοιμαστούν. Αυτά όμως, αυτές οι δεξιότητες δεν περιέχονται σε κανένα από τα βιογραφικά ή τέλο πάντων ή στην ύλη ε, οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτά θα πρέπει να προσέξουμε ως προβλήματα. Επίσης, νέα τομέα, νέα θέματα. Τα προβλήματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με την εργασία στην ψηφιακή τεχνολογία. Και δεν είναι μόνο σωματική υγεία, είναι και το στρες. Νευρολογικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, επιπτώσεις από τέτοιου είδους εργασία. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθούν, να αντιμετωπιστούν. Οπότε δύσκολο και να θεσπίσει κανείς κάποια πρότυπα. Άρα θα πρέπει και αυτά να τα προσέξουμε και να τα αναδείξουμε στην γνωμοδότηση. Είναι σύντομη αυτή η γνωμοδότηση και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι δυναμικά θα κινηθούν να προτείνουν τροπολογίες και έτσι να ε, προωθήσουν κάποιες ιδέες που έχουν προκύψει από τις συζητήσεις μας εδώ στην Επιτροπή και το αποτέλεσμα να είναι αξιόλογο. Θα γίνει αξιόλογη συζήτηση και οι προθεσμοί για τις ε, τροπολογίες πιέζει. Είναι σύντομη. Είναι 31 Ιανουαρίου. Θα τα πούμε την Τρίτη στο επόμενο Στρασβούργο. 14 Φεβρουαρίου. Επίσης, για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, οπότε να είμαστε έτοιμοι για να κατεβάσουμε αυτή την γνωμοδότηση ε, στην Επιτροπή την ε, τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου. Ευχαριστώ κύριε Λαουρίστη, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να είναι εδώ ο συγητής του ΕΛΚ. Α, εδώ είστε. Ε, κυρία Γεσλοβιέκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο Κύριε Σέτμαν είναι σκιώδης εισηγητής, δυστυχώς όμως δεν μπορούσε να έρθει. Γι' αυτό θα τον αντικαταστήσω και θα παρουσιάσω αυτά που θα ήθελε να πει. Η εκβιομηχάνηση της... Η ψηφιοποίηση μάλλον της βιομηχανίας έχει πολλές... Έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Το 2015 είδαμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπρόσθετα κέρδη 150 δισεκατομμύριων ευρώ ε, με την ψηφιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ θετικό για την ε, οικονομία μας. Ωστόσο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και εμπόδια τα οποία καθιστούν αδύνατο να ε, εκμεταλλευτούμε το πλήρες δυναμικό πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι της άποψης ότι ε, υπάρχουν πολλά, πολλές φορές ανυπέρβλητα, εμπόδια και περίπου το ίμιση των εργαζομένων θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετά προσόντα για να ανταπεξέλθουν στην σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Η λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και θεωρώ ότι οι διαφορές ανάμεσα σε εμά και τις Ηνωμένε Πολιτείε θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Το περασμένο έτος ο συνάδελφος κύριος Χέτμαν ήταν παρόν σε ένα σεμινάριο στο οποίο Έγινε μια σύγκριση της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας από την άποψη της νοοτροπίας και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πάρει στα σοβαρά την ψηφιοποίηση, την ανάγκη γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως πρέπει οι ίδιοι πρώτα να αλλάξουμε νοοτροπία έτσι ώστε να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιοποίηση. Γι' αυτό χρειάζεται η απόκτηση πρόσθετων προσόντων και οι εργαζόμενοι πρέπει λοιπόν να δείξουν ευελιξία έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και τις δεξιότητές τους. Η ψηφιοποίηση λοιπόν της βιομηχανίας θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι που αφορά και τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν ε, αρμοδιότητα όλων. Αποτελούν κομμάτι των ε, soft skills, των ήπιων λοιπόν δεξιοτήτων. Κάτι το οποίο πιστεύω πως θα έπρεπε να αρχίσει να καλλιεργείται ήδη από το δημοτικό. Διότι η έλλειψη δεξιοτήτων ψηφιακών νομίζω πως αποτελεί κίνδυνο για την ε, περαιτέρω εξέλιξη της ε, αγοράς εργασίας. Ο συνάδελφος ε, έχει κάποιες σχετικές τροπολογίες, τις οποίες θα υποβάλει και αφορούν ακριβώς αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Ζλωτόφσκι εκ μέρους της ομάδας ECR. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το κείμενο αυτό. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν περιορίζεται μόνο στην ε, απαρίθμηση των ε, πλεονεκτημάτων της ψηφιακής οικονομίας. Νομίζω ότι χρειάζεται μια θεμελιώδης ε, αλλαγή νοοτροπία. Πρέπει να δούμε όχι μόνο τα πλεονεκτήματα αλλά και τι απειλές που έρχονται μαζί με την ψηφιοποίηση της ε, βιομηχανίας. Η ψηφιακή επανάσταση λοιπόν δεν μας παρέχει μόνο νέα μέσα επικοινωνίας, νέα μέσα ε, διασκέδασης αλλά και οικονομικού τύπου δυνατότητες και ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σαφές πως χρειάζονται και ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί μόνο σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο δηλαδή στη δευτεροβάθμια και ε, μετέπειτα εκπαίδευση, αλλά ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει κάποιος νωρίς. Επίσης, είναι πολύ σημαντική και η κατάρτιση και η μετεκπαίδευση των εργαζόμενων. Κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο αποκλεισμό από τις ψηφιακέ δεξιότητες οδηγεί και σε αποκλεισμό πάρα πολλών ε, ανθρώπων από την αγορά εργασίας. Και αυτό οδηγεί και σε κενά μετά στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν αυτά τα κενά, να καλυφθεί ε, αυτή η έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες και πρέπει λοιπόν, θεωρώ, να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα που μας δίνουν ορισμένες εταιρείες ε, και να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Βλέπουμε ότι στον τομέα του τουρισμού έχουν γίνει πάρα ε, πολλά και έχει εξυγχρονιστεί ακριβώς λόγω της ψηφιοποίησης. Μετά, χρειάζεται φυσικά ένας μηχανισμός προστασίας που θα συμμορφώνεται με τους υφιστάμενους κανόνες και γι' αυτό χρειάζεται ευελιξία στη διοίκηση και χρειάζονται και κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Ε, και φυσικά χωρίς να ξεχνάμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δικαίωμα, για παράδειγμα, ε, στην ανάπαυση, σε άδεια κτλ. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ε, στα εργαλειοθήκη μας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αξιοποιήσουμε την τηλεργασία διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και όσοι, για παράδειγμα, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά να μεγαλώσουν και δεν μπορούν να βρίσκονται με φυσική τους παρουσία ε, σε κάποιο κέντρο κατάρτισης. Επίσης, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντική και εδώ βλέπουμε τεράστια διαφορά ανάμεσα στις πόλεις και την Ήπεθρο. Είναι λοιπόν ε, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς, η οποία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με επενδύσεις. Οι επενδυτές θέλουν όμως και εκείνοι ερεθίσματα έτσι ώστε να ε, δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και όλα αυτά που σας ανέφερα θα τα ε, δείτε και γραπτός με τη μορφή τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελεύθερους θα πάρει το λόγο ο Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και την εισηγήτρια την κυρία Λαόρεστη για το προσχέδιο ονομοδότησης, και οποίο του καλωσορίζω. Είμαι νέος, νέο μέλος της Επιτροπής και είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με το θέμα, επομένω θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη αν επαναλάβω κάτι. Η ψηφιακή οικονομία έχει μια τεράστια δυναμική μεταμορφώσεις, μετασχηματισμού της αγοράς, της, των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Βεβαίως δημιουργεί και προκλήσεις, κυρίως στη σχέση με την οργάνωση της εργασίας. Δεν το παραγνωρίζω αυτό. Όμως εμείς ως φιλελεύθεροι ξεκινούμε ε, σκεπτόμενοι ότι αυτές οι αλλαγές ανοίγουν ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Στη χώρα μου διαπιστώνουμε πώς αυτή η ψηφιακή οικονομία έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι καιρό είναι να βοηθήσουμε τον, την βιομηχανία να βρεθεί ο ίδιος, να, να, αναλάβει πρωτοβουλίες ο ίδιος ο τομέα της βιομηχανίας στην ψηφιακή οικονομία και να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορούμε να αναμένουμε τη δημιουργία 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020 μόνο μέσω των startup. Θα Ήθελα επίσης να κάνω παρατηρήσεις και θα κάνουμε και προτάσεις οι οποίες θα κατατείνουν προς μια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση. Ε, εμείς έχουμε αμφιβολία όσον αφορά την αρχή της πλήρους πρόσβασης στο γρήγορο ίντερνετ. Αυτό είναι ίσως υπερβολικά φιλόδοξος στόχος και καλύτερα να θέσουμε έναν πιο, πιο ρεαλιστικό. Το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι συνέπειες του βεβαίως θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει, αλλά μόνο όταν αυτό το πλαίσιο δημιουργεί αρνητικές συνέπειες. Αντιθέτως, όταν η ψηφιοποίηση της, αγορά, της οικονομίας έχει θετικές επιπτώσεις, θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Πέντε παράγραφος, πέμπτη παράγραφος. Όπως έχει διατυπωθεί, δεν μπορώ να την ε, δεχτώ. Η Σουηδία, η χώρα μου, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η εξάλληψη των ρυθμιστικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις έχει βοηθήσει τον τομέα της τεχνολογίας. Ξαναλέω, δεν παραγνωρίζω τα προβλήματα, δεν κλείνω τα μάτια μου σε αυτά, αλλά λέω ότι υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Γι' αυτό νομίζω και αυτό είναι σημαντικό κατά την απόψή μου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στα ζητήματα του συλλογικών διαπραγματεύσεων, του δικαιώματος της απεργίας, του δικαιώματος του συναφρίζεστε. Αυτά είναι δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να... τα οποία είναι πολύ σημαντικά τα προασπίζεται αυτός που μπορεί να τα επιβάλλει. Ο εγγυητής αυτών των δικαιωμάτων είναι μόνο εκείνος που έχει την εξουσία να τα εξασφαλίζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας. Ακόμα λοιπόν και για μας στην Άλτε που είμαστε πάντα υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωση, πάντα ίσω υπερβολικά υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωση και Αμερικού, θεωρούμε ότι είναι δικαιώματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε, ε, να, τα υπερασπιστεί το κράτος. Η ευελιξία, η τηλεεργασία, η κινητικότητα και αυτές δίνουν ευκαιρίες και θα πρέπει να βρούμε ε, έναν τρόπο να δείξουμε ότι αυτό, αυτές οι τάσεις δεν δημιουργούν μόνο προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Δηλαδή ότι υπάρχουν και δύο πλευρές. Κλείνω λέγοντα ότι θα υποβάλω ορισμένες θα υποβάλουμε ορισμένε τροπολογίε έτσι ώστε να εκφράσουμε αυτά που σας ήδη, ήδη σας περιέγραψα, τις θέσεις δηλαδή της άλλης, τι ονομοδότης της ηγετρίας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόπες Περμέιρο που την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς η εργατική νομοθεσία καλύπτει ε, την ψηφική τεχνολογία. Άρα πρέπει να γίνει ανάλυση όσον το χρόνο εργασίας και επίσης τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων. Τώρα αποκρύπτεται η εξάρτηση των εργαζομένων. Ασφάλεια και υγεία στον χώρο της ε, εργασίας. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η απεργία, όπως το δικαίωμα στην συλλογική σύμβαση. Άρα θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο και να προβληματιστούμε για το μέλλον της απασχόλησης, για την κατανομή της εργασίας, αλλά και την εκπαίδευση στα ψηφιακά. Εν τέλει να σας πω ότι οι προτάσεις της κυρίας Λαουρίστην όπως και η αναγνώριση από πλευράς της των κοινωνικών εταίρων πάνε προς την σωστή κατεύθυνση και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες πιστεύω ότι παραγωγικά πρόκειται να συνεργαστούμε και, και τις τροπολογίες μας. The is by Ποιος εκπροσωπεί τους πράσινους. Κανείς. Δεν παρευρίσκεται λοιπόν κάποιος εκπρόσωπος ούτε από το EFTD, ούτε από την ENF. Και άρα ποιος, σε ποιον θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Η κυρία Λοβέκα. Δεν σας είχα δει. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα αυτό. Μια και αφορά την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά επίπεδα ψηφιοποίησης και για να αποτρέψουμε αυτήν την ε, δυστοπική πρόβλεψη που, είπε, που αναφέρει η συνάδελφος με το 40% των επαγγελμάτων που κινδυνεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να δώσουμε μία ευκαιρία στο σύνολο της Ένωσης θα πρέπει καταρχάς να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα που απειλούνται από την ψηφιοποίηση. Και να είμαστε σαφείς, να ορίσουμε και τους ε, επιμέρους παράγοντες, να ονομάσουμε ακριβώς ε, ποιος κινδυνεύει. Πρέπει όμως επίσης να χρησιμοποιήσουμε και την ψηφιοποίηση. Και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει και μία μελέτη έτσι ώστε να δούμε όχι μόνο ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την ψηφιοποίηση αλλά και ποια θα ωφεληθούν περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν ε, μέσα στη διάθεσή μας διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν γι' αυτό, έτσι ώστε να αποφύγουμε το τσουνάμι της ψηφιοποίησης με τις, και τις αρνητικές του συνέπειες. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε το θέμα πολύ στα σοβαρά όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θεωρώ πως πρέπει η ε, ψηφιακή εκπαίδευση να αρχίσει ήδη από την, ε, από την σχολική ηλικία, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε οι νέοι να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο, εάν το επιθυμεί, αν έχετε κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε κάποια πρόσθετα σχόλια. Σημειώσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα ακούστηκαν και ε, θα ε, ήθελα να πω ότι συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάουριστιν, θα θέλατε να κάνετε κάποια τελευταία σχόλια. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και εισηγητές και ε, όσους ενδιαφέρθηκαν και συνεργάστηκαν μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να συνεισφέρει τα μέγιστα. Να απαντήσω ίσως στην, στον συγητή των φιλελεύθερων για την καθολική πρόσβαση. Ε, να σας πω ότι στη δική μου χώρα, την Εστονία, οι Σουηδικές τράπεζες έκαναν μια μεγάλη συνεισφορά προς αυτήν την καθολική πρόσβαση, διότι Έγινε ρευστοποίηση των υποκαταστημάτων στα μικρά χωριά. Έκλεισαν τα υποκαταστήματα λοιπόν στα χωριά της Εστονίας διότι δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης αυτών και ως αποτέλεσμα αυτού ακόμα και στα μικρότερα χωριά άρχισαν όλοι να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές ε, τραπεζικές υπηρεσίες για τις συναλλαγές τους. Και μάλιστα προσφέρθηκαν μαθήματα χρήσης του διαδικτύου σε 100.000 ανθρώπους ηλικιωμένους. Είναι λοιπόν βασική η καθολική πρόσβαση στην ψηφιοποίηση, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για νέα ψηφιακή αγορά και να αποκλείουμε ορισμένους ε, ανθρώπους, κάποιες μερίδες του πληθυσμού, διότι αυτοί είναι επίσης και πιθανοί πελάτες των ψηφιακών επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονιστεί ότι οι ψηφιακές υποδομές πρέπει να βρίσκονται παντού και στο μικρότερο χωριό ακόμα. Αυτό είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έγγραφο της Επιτροπής είναι μια υπόσχεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δικό μας έργο είναι να δούμε πώς μπορούμε να παροτρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και με ενδιαφέρει πολύ ο τομέας της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τι δουλειά μπορεί να κάνει μετά, οι θέσεις απασχόλησης, αν θα χαθούν, αν θα δημιουργηθούν και άλλες, να πω ότι οι μελέτες δείχνουν ότι, για τη ότι από μία τέτοια ε, θέση απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων δημιουργούνται άλλες πέντε. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι όντως κινδυνεύουν να χαθούν κάποιες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν περισσότερες. Ας μην φοβόμαστε λοιπόν την αλλαγή, την ψηφιακή αλλαγή. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την ανταλλαγή απόψεων. Σας περιμένω στο Στρασβούργο στις 14 Φεβρουαρίου για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ελπίζω να έχω μέχρι τις 31 Ιανουαρίου πολλές ενδιαφέρουσες και περιεκτικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίε είναι 31 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε 22 με 23 Μαρτίου. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δημιουργία ενός κοινού ε, πλαισίου... Πλαίσιο για ευρωπαϊκές θεστικές για πρόσωπα και και νοικοκυριά με στοιχεία από δείγμα ατομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να δούμε το πώς θα μπορέσουμε How we can, Εδώ πέρα πώς θα έχουμε στοιχεία από διαφορετικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο για ε, το μέλλον και για τόσα γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μέσετς που είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω ότι όπου να είναι θα έρθουν οι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μπορέσουμε να υποβάλουμε τα απαντήσει. Να ακούσουμε και την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά το σχετικό νομοθέτημα. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για τεχνικό κανονισμό και τίποτε άλλο. Όμως αυτό δεν ισχύει. Δεν το λέω αυτό γιατί είμαι ο συντάκτης και θεωρώ σημαντικό το θέμα μου, αλλά γιατί θεωρώ, όπως λέει και το προήμιο του κανονισμού, ότι αν συμφωνήσουμε με το ότι όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ενημερωμένα και συγκρίσιμα δεδομένα. Κάνει ό,τι μπορεί η Eurostat για τέτοια δεδομένα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Η συλλογή των δεδομένων με τις έρευνες είναι γνωστό ότι έχει προβλήματα ή θα πρέπει κανείς να έχει συγκεκριμένα δεδομένα ή κανείς μπορεί να έχει αξιόπιστα δεδομένα ή να έχει ενημερωμένα. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να συμβιβαστεί, να συμβιβαστεί όσον αφορά την ποιότητα και την συγκριτικότητα για την άλλη μεριά να έχει επικαιροποιημένα. Άρα γι' αυτό το έχουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό είναι θέμα πολιτικής άρα δεν είναι θέμα τεχνικό. Άρα θα πρέπει να δούμε το πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται μία έρευνα. Ε, αυτό δεν είναι ζήτημα του πότε θα τα καταφέρει καλύτερα η κάθε εταιρεία ή η κάθε υπηρεσία τέλο πάντων, η κάθε στατιστική υπηρεσία κράτου μέλου σε συνεργασία με την Eurostat. Το θέμα είναι τι πολιτική θα ασκήσει κανεί, ώστε να έχουμε επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στοιχεία. Είναι υψηλό στι λεπτομέρειε, γιατί δεν μπορώ τώρα να σα παρουσιάσω το σχέδιο κειμένου. Ε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά είπαμε ότι πρόκειται για κανονισμό πλαίσιο που θα καλύψει τους επόμενους κανονισμούς που θα ακολουθήσουν για αυτό το θέμα. Μέσα σε πέντε χρόνια πιστεύω θα έχουν καλυφθεί οι έρευνες των δεδομένων από τέτοιους κανονισμού. Θα είναι το πρώτο βήμα δηλαδή αυτό ο εικονισμό. Οπότε παρακαλώ ποιο ενδιαφέρεται και οι ηγητές να δραστηριοποιηθούν γιατί ήρθε η ώρα να προτείνετε τι. ιδέε σα. Βέβαια ξέρουμε ότι έχουμε περιορισμό ε, και κυρίω οικονομικό περιορισμό. Βέβαια εγώ ω ηγητής θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για όλου σα και να δούμε πώ θα βελτιώσουμε την ε, ποιότητα των δεδομένων με τον κανονισμό και επίσης να δω το πώς θα μπορέσουμε να μείνουμε μέσα στα οικονομικά ή δημοσιονομικά πλαίσια που υπάρχουν. Και είναι σημαντικός αυτός ο περιορισμός. Όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με κοινωνικέ επιστήμε, όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για τέτοιου δεδομένα, γνωρίζουμε ότι τελικά το κοινωνικό κόστο να προσπαθεί κανένα να έχει συγκρισιμότητα δεδομένων ε, στο τέλος ξέρει ότι αν από την αρχή βγήκε ο κανονισμός τότε θα ήταν πράγματα καλύτερα. Επομένω, η συγκρισιμότητα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Αλλά και αυτό απασχολεί και τους χρήστες των δεδομένων και όχι μόνο τους κοινωνικούς επιστήμονες. Όλους τους εμπλεκομένους, όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους και η συγκρισιμότητα των δεδομένων μέσω των ε, καλύτερων ερευνών. Τώρα, κάτι άλλο σημαντικό. Έχουμε κάποιο διαχωρισμό. Κατανομή, διαχωρισμό, πώς το πούμε, τόσο να δεν είναι το ίδιο έρευνες. Θα ήθελα να ρυθμίσουμε σε κάθε επίπεδο τα δεδομένα. για όλους του τομεί κοινωνική πολιτική. Γιατί θα έρθουν να κάνουν ε, οι χρήστες ε, σύγκριση δεδομένων μεταξύ ας πούμε Γερμανίας και Λουξεμβούργου. Και αν δεν έχουμε φροντίσει όλα τα επίπεδα σύγκριση δεδομένων, δεν έχει νόημα τότε μετά για το χρήστη η δουλειά μας. Είναι κοινό μας ο στόχος μόνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, Περιμένω πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και με την Επιτροπή και με τους συναδέλφους. Για να δούμε πώς θα είναι ο κανονισμό, πόσο ενδελεχής θα είναι. Και να δούμε τι θα γίνει με τις εφαρμοστικές πράξεις ή τις κατανάθεση κατεξιοδότηση πράξης. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, το πώς θα γίνει. Το συζητήσουμε με τους κοιοδησηγητές και μετά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω τελικά και με το Συμβούλιο. Αυτά. Σαν εισαγωγή από μένα. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Uh, Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις πολιτικές ομάδες έχει δείξει το ενδιαφέρον που πρέπει με την παρουσία της αυτήν εδώ τη συζήτηση. Βέβαια, αρχίσαμε και 15 λεπτά νωρίτερα, οπότε αυτό ίσως σημαίνει ότι σε 15 λεπτά θα φτάσουν μέλη γεμάτα ενέργεια και όρεξη για συζήτηση. Και πάνω απ' όλα με μαχητικό πνεύμα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να δώσω ακόμα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και να πω ότι νομίζω εννέα ή 10 μήνες πριν είχαμε ξανασυναντηθεί για το ίδιο θέμα και ήταν πολύ έντονη η συζήτηση παρά το αργό της ώρας. Και οι ευρωβουλευτές άφησαν να εννοηθεί ότι ήθελαν πολύ να ξανασυναντηθούν με την Κομισιόν τουλάχιστον άλλη μία φορά για να συζητήσουν το θέμα. Και ελπίζω να φτάσουν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές σύντομα. Έχω εδώ έναν κατάλογο σκιωδών εισηγητών, αλλά πολλοί από αυτούς λείπουν επειδή δεν τους επιτρέπει το πρόγραμμα να έρθουν. Θα ήθελα λοιπόν να τους περιμένουμε και μέχρι τη στιγμή που θα έρθουν νομίζω πως θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λάουριστέιν από την Εστονία, η οποία γνωρίζει ακριβώς όλα τα προβλήματα που υπάρχουν πίσω από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι κατάλληλη ευκαιρία και πράγματι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Με τα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα, νομίζω πως μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ε, εξή προσεγγίσεις. Καταρχάς, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εθνικές ε, στατιστικές, τα στοιχεία. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον ε, ορισμό τους και εάν υπάρξει κάποια εναρμόνιση στα εθνικά στατιστικά στοιχεία, τότε θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικονομικά να κάνουμε σύγκριση για πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έπειτα, πρέπει να γίνονται μελέτες, να δούμε τις ε, πανευρωπαϊκές μελέτες, μελέτες στα νοικοκυριά. Ε, αυτό δεν είναι υπεύθυνη η Eurostat, αλλά η ESS, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Στατιστική Υπηρεσία. Χρειάζεται όμως χρηματοδότηση. Και έχει πέσει θύμα απώλειας κονδυλίων από πολλά κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Καταρχάς δημιουργώντα μια καλύτερη Eurostat, μια Eurostat η οποία υποχρηματοδοτείται. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διαφυλάξουμε την ε, συνοχή σε βάθος χρόνου. Εάν καταφέρουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό, θα ωφελήσει όχι μόνο αυτόν τον τομέα της ε, πολιτικής, αλλά και γενικότερα τις κοινωνικές επιστήμες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη εισέλθει στην εποχή των ε, big data. Αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων, λοιπόν, πρέπει να μας βρει έτοιμους σε όλους τους τομείς και στις κοινωνικές επιστήμες, διότι δεν έχουν γίνει ακόμα τα βήματα που πρέπει στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που στο σχόλιο σας συμπεριλάβατε και την ψηφιοποίηση, θέμα που μόλις συζητήθηκε. Κύριε Πυρίνσκι, αρχίσαμε ήδη, γιατί αρχίσαμε νωρίτερα. Ο κύριος Μέσαριτς είμαι σίγουρη πως θα επιστρέψει για να τοποθετηθεί. Ήδη έγινε μια πρώτη παρέμβαση. Θα δώσω τώρα σε εσά το λόγο, σύμφωνα με τον κατάλογο των ομιλητών που έχω μπροστά μου. Κύριε Πυρίνσκι, λοιπόν, εκ μέρου τη ομάδα SND. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι το θέμα αυτό είναι ζωτική σημασία και εξίσου σημαντική είναι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα καθορίσει την έκταση την οποία θα λάβουν τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Φυσικά και η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική και επίσης θα μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κοινωνική μας πολιτική. Νομίζω πως η Επίτροπος Τάισεν έχει αναφερθεί πολύ εύστοχα σε αυτό, σε, στο παρελθόν. Χρειάζεται να βελτιωθεί η ποιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Και η ίδια η Επίτροπος βάζει την ε, κοινωνική, το βάζει αυτό στο κέντρο της ε, κοινωνικής ατζέντας του τριπλού Αλφα. διότι είναι το μέσο με το οποίο θα επιτύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσες πολλές διαφορετικές προτάσεις υπό ένα πλαίσιο. Αυτές τις ασκήσεις, αν θέλετε, που θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη, πιο φιλόδοξη ίσως προσέγγιση. Η οποία βέβαια δεν έρχεται χωρίς κινδύνους. Μία τόσο ριζική μεταρρύθμιση έχει κινδύνους και ο μεγαλύτερος όπως ε, έχει αναφερθεί είναι ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε μείωση της... του χρόνου ο οποίος χρειάζεται για να συλλεχθούν και να παρουσιαστούν αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα λοιπόν, αυτά τα στατιστικά στοιχεία έπρεπε να είναι έτοιμα ένα χρόνο προτού αρχίσει η επεξεργασία τους. Και αυτές ε, λοιπόν οι μελέτες που μπορείτε να φανταστείτε ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Χρειάζεται... Ε, χρειάστηκε λοιπόν πολλές φορές να μειωθεί ο χρόνος στους 11 μόλις μήνες. Και αυτό θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε ένα χρόνο. έτσι ώστε να τον αφιερώσουμε σε άλλες ενέργειες. Τώρα δεν θα κρίνω κατά πόσο αυτό βελτιώνει την κατάσταση. Υπάρχουν ορισμένοι δείκτες σχετικά αν ενδιαφέρεστε. Και δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα του να κόψουμε χρόνο Τώρα, πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει και ότι αυτός ο νέος τρόπος συλλογής δεδομένων θα δώσει περισσότερη ευελιξία. Ακριβώς γιατί αυτός ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών, οι τάσεις που παρατηρούνται κτλ μεταβάλλονται ταχύτατα και με τρόπο ε, μη αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, χρειάζεται να συλλέγονται δεδομένα ε, πιο γενικά, πιο ευρύτερα και φυσικά χρειάζεται και αντίστοιχη μεταβολή των βάσεων δεδομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική, εδώ θα παρουσιαστούν ίσως κάποια προβλήματα για να επιτύχουμε αυτή την ευελιξία. Θα ανέβει και το κόστος, θα αυξηθούν οι δαπάνες και τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν και την ετοιμότητα και την δυνατότητα να απορροφήσουν αυτό το πρόσθετο κόστος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, όπως και δίποτε. Και χρειάζεται δέσμευση, χρειάζεται φιλοδοξία και ετοιμότητα από τα κρατη για να αρχίσουν την εφαρμογή αυτής της άσκησης. Και πάνω απ' όλα σκληρή και εντατική δουλειά. Γιατί υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, υπάρχει διαφορά στον όγκο των δεδομένων και ας μην ξεχνάμε πως και οι μελέτες είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτάξει και άλλο ένα βασικό επιχείρημα, ότι δηλαδή όλο αυτό θα επιφέρει μια συνοχή. Θα υπάρχει μεγαλύτερη οριζόντια σύγκληση και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα η τα ευρήματα να συνδυαστούν για να οδηγήσουν σε καλύτερη ενημέρωση προτού ληφθούν αποφάσεις. Προς το παρόν, ε, αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία συναντούν δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες έχουν, για παράδειγμα, να κάνουν με τη μέτρηση της ανεργίας, με ε, τη μέτρηση της ανεργίας σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτό λοιπόν χρειάζεται διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζονται σαφείς οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τώρα κάτι γενικότερο Νομίζω πως αναφέρθηκε ήδη από την Κομισιόν πως αυτά τα κοινωνικού χαρακτήρα δεδομένα είναι λυπή. Υπάρχει και ε, ένας άλλος μεγάλος όγκος δεδομένων που αφορά τη... τα στατιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων δομή των κερδών, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Υπάρχουν σχετικές μελέτες και νομίζω πως τα ευρήματα αυτών των μελετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής. πρωτού μπούμε σε λεπτομέρειες και δούμε ε, ακριβώς το τι σημαίνει η πρόταση σε αυτό επίπεδο. Ενδεχομένως να πλέουμε σε χαρτογράφητα νερά, αλλά αν μας διακρίνει η αντικειμενικότητα και προσπαθήσουμε όντως να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στην άσκηση αυτή, θα δούμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. You didn't hear the ε, δεν είχατε ακούσει λοιπόν την τελευταία μου παραβίση. Έλεγα ότι η πρόσωπο τη κυρία, της Άλτε δεν είναι εδώ, αλλά και η Λίν Μπόιλ είναι εδώ και θα τη δώσω το μέσο στο λόγο. Ευχαριστώ. Έχω διάφορα θέματα για το, στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με το ζήτημα που συζητούμε. Στόχος ε, αυτού του κανονισμού είναι να οργανωθεί καλύτερα ο τρόπος συλλογής στατιστικών στοιχείων, στοιχεία που συλλέγονται για την χάραξη πολιτικών και τα οποία χρησιμοποιούνται και ε, ωφελούν όλα τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η ανεργία, η φτώχεια, η κινητικότητα, η εκπαίδευση κτλ. Για να λαμβάνουμε, να χαράσουμε πολιτικέ, να λαμβάνουμε αποφάσεις στα θέματα αυτά, χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοιχεία. Επομένως, πιστεύω ότι πράγματι ε, θα βελτιωθεί η ευημερία των πολιτών μας ε, και από οικονομικής πλευράς και από κοινωνικής πλευράς αν πετύχουμε τους στόχους που θέτει αυτός ο κανονισμός. Όπως λοιπόν σωστά είπε ο εισηγητής, αυτή η πρόταση κανονισμού είναι πολιτική, δεν είναι απλώς τεχνική. Έχουμε διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Φαίνεται πλέον ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων μπορεί να γίνει με τρόπο πιο ε, ευέλικτο και πιο φιλικό προς τον χρήστη. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ε, για να καταλάβουμε καλύτερα πώς θα λειτουργεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις συνθήκες διαβίωσης και επίσης πώς θα περάσουμε από την, κάθε, την, την περιοδικότητα κάθε τέσσερις, ε, τέσσερις φορές το χρόνο στην περιοδικότητα κάθε έξι φορές το χρόνο ε, χωρίς αυτό να προκαλέσει προβλήματα και να υπονομεύσει τον κύριο στόχο του κανονισμού. Χαίρομαι που θα ε, υπάρχουν πλέον, θα συλλέγονται πλέον και στατιστικά στοιχεία για τον, τον πλούτο είναι απαραίτητο αυτό, κατά την άποψή μου, για να γνωρίζουμε ποια είναι η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3. Θα ήθελα να ε, μάθω όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει οικονομική βοήθεια στα κράτη-μέλη, μάλιστα δεδομένου ότι ορισμένε από αυτέ τι ε, μελέτε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων θα είναι υποχρεωτικέ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον κανονισμό αυτό ε, φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ε, πιο συγκεκριμένα ε, μελέτες, δείκτες και στατιστικά στοιχεία που θα απαιτείται από τα κράτη-μέλη να αποστέλουν στην Eurostat. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ο κανονισμός πηγαίνει προς μια σωστή κατεύθυνση, Ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την διάθεση να συζητήσει μαζί μας για τα ζητήματα που μας απασχολούν και τις ανησυχίες που έχουμε με αυτόν τον κανονισμό, μαζί με τα κράτη-μέλη φυσικά και φυσικά και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος από τους πράσινους, από την EFTD. Δεν έχει ορίσει καν. Σκιώδη. Ε, ο κύριο Μαχτάν, μήπω θα ήθελε να εκπροσωπήσει του ΙΕΝΕΦ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η αρχική ιδέα, δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τα στατιστικά στοιχεία για στο κοινωνικό επίπεδο, το οποίο να είναι επικαιροποιημένο και αξιόπιστο, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ωστόσο, Έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία και πολλές ανησυχίες για τα στατιστικά στοιχεία όταν μιλούμε για απλοποίηση των εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα όργανο το οποίο δεν είναι εκλεγμένο, θα έχει τη δυνατότητα μέσω πράσιων κάτι εξουσιοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού που μας προτείνει, να τροποποιεί τα στατιστικά στοιχεία που θα προβλέπεται να συλλέγονται. Εδώ τίθενται πολλά ζητήματα. Αν έχουμε διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας, αυτό θα οδηγήσει σε διαφορετική μοντελοποίηση και σε διαφορετική συμπεράσματα. Επίσης, ζητείτε να αποστέλλονται ε, στατιστικά στοιχεία και αρχεία με στατιστικά στοιχεία που είναι στο, κέντρο της λειτουργίας της, της διοίκησης κάθε κράτους και αυτό επίσης μας ανησυχεί. Λέγεται από, στον κανονισμό, στην, στο σημείο σημείωμα, ότι αυτή η προσπάθεια θα βοηθήσει και στο σχέδιο μέχρι το 2020 στην καλύτερη λειτουργία της Ευρωζώνης και σε μια σειρά σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες όμως όλες έχουν, αυτές έχουν αποτύχει επανειλημμένος. Σας ευχαριστούμε κυρίως Μέτσερνιχ ε, από τους πράσινους είχατε λάβει το λόγο και προηγουμένως αλλά δεν ήταν εδώ οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν μιλήσατε πως θέλετε να ξαναπείτε αυτά που είπατε πριν δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλετε Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο, λέει ο κύριο Ευχαριστώ για όλε τι παρεμβάσει. Ήδη φαίνεται ότι θα αποδώσει καρπού η ανταλλαγή απόψε με του κοιότε ηγητέ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πολύ το θέμα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να εξαθέσει κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ακούσαμε αυτό ήδη από όσους μίλησαν. Να δούμε επομένω του αρχικού στόχου, να δούμε σε τι πλαίσια κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ήθελα να σας πω κάτι, αφού ήδη έχω τις με κάποιους υπαλλήλους της Κομισιόν. Ο κανονισμός αυτός έχει εξαντλητικά συζητηθεί με τις θεσχές υπηρεσίες των κρατών μελών. Βεβαιώστε παρακαλώ. Ότι αυτό έχει γίνει και δεν χρειάζεται να το κάνουμε αργότερα. Τώρα αυτό που κυρίως με απασχολεί σε αυτή τη φάση είναι το εξή. Το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τα όρια των τεχνικών θεμάτων και τα όρια και τη διάκριση με τα πολιτικά. Έτσι δεν διαμορφώσουμε την πρότασή μας. Ρώσο από την αριστερά. Τι θα γίνει, πώς η κατεξιδότηση πράξης ε, πρόκειται να λειτουργήσουν. Όπω σα είπα διαμορφώνεται η πρότασή μας, οπότε τώρα δεν μπορώ να σα πω περισσότερο για το σχέδιο κειμένου. Πάντως, συμφωνώ με το στόχο που έχετε τάξει και όπως και οι συνάδελφοι θεωρώ ότι είναι σημαντική υπόθεση. Άρα, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη δουλειά μας. Thank you. Then I'll give the floor to uh, uh, perhaps Galo Guay uh, the Director of Social Statistics. δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Διεθνή Στατιστικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω και ο λόγος του κανονισμού είναι, όπως προαναφέρθηκε, το να έχουμε ε, ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία και αξιόπιστα ευρωπαϊκές πολιτικές, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, την κοινωνική ατζέντα, την Ευρώπη 2020 κλπ. Οπότε, εμείς έχουμε όλο ένα και περισσότερη ζήτηση για πολλά θέματα και περιφερειακά και εθνικά ε, ανάπτυξη, απασχόληση ε, ανισότητες, κοινωνική περιθωριοποίηση ε, παιδεία, δεξιότητες ψηφιακέ δεξιότητε, κοινωνική πρόνοια, ευημερία. Οπότε και θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση με ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία και αξιόπιστα. Οπότε επί κάποια χρόνια συνεργαζόμαστε με τις αισθητικές υπηρεσίες των κρατών μελών για να δούμε πώς θα εξυγχρονίσουμε αυτά τα κοινωνικά στατιστικά στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στι ανάγκες Some Να σας πω τι γίνεται ανάλογα με αυτά που και εσείς δείξατε. Πρώτα πρώτα, το σχέδιο κανονισμού σήμερα συζητάμε είναι ο πρώτος κανονικός πλαίσιο γιατί έχουμε τρεις συνεργασμούς ο, ο πρώτος αφορά τις Έλληνες, ο δεύτερος αφορά τον ε, πληθυσμό και τις ε, απογραφές και θα υπάρξει και ένας τρίτος κανόνας πλαίσιο ακόμα πιο μετά που θα αφορά τα δεδομένα για διοικητικά θέματα. Παιδεία, και κοινωνική πρόνοια. Προχωρήσαμε λοιπόν βήμα-βήμα για να είμαστε πιο πρακτικοί. Όλα αυτά συναρτώνονται μεταξύ τους για να υπάρχει συνέπεια και τελικά πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια σφαιρική πλήρη θεστική βάση. Ξεκινήσαμε με τις έρευνες γιατί θεωρούμε ότι από πλευράς ε, ολοκληρώσεις, κωδικοποίησης, βελτίωσης έτσι πρέπει να γίνει. Να σας δώσω επίσης και κάτι άλλο. Αυτός ο κανονισμός απλουστεύει γιατί εδώ θα συγκεράσουμε σε ένα πλαίσιο διάφορες συλλογές δεδομένων. Θεωρούμε ότι θα έχουμε τώρα πιο πλήρη δεδομένα, πιο πλούσια. Υπάρχει χώρος στις έρευνες. Υπάρχουν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ερευνών. Και έτσι θα καλύψουμε πολυδιάστατα φαινόμενα όπως τις δεξιότητες. για τις δεξιότητες, για την παιδεία και όλα αυτά θα αξιοποιηθούν από τις πολιτικές όποτε χρειάζονται πληροφορίες για να μπορέσει κανείς να καταλάβει την κατανάλωση αλλά και τον πλούτο. Τώρα, τα χρονικά όρια, τα χρονικά πλαίσια. Μετά την περίοδο αναφορά έχουμε μία τριετία. Δύο, δύο, δύο για αυτό είναι ο Δύο μετά την περίοδο αναφορά. Οπότε και θέλουμε ε, δραστικά να βελτιώσουμε αυτά τα πλαίσια κατά ένα χρόνο. Οπότε αυτά τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα όταν ξεκινά το ευρωπαϊκό εξάμεινο και έτσι να εξυπηρετούν το εξάμεινο. Επίσης, ξέρουμε ότι αυτές οι εξελίξεις κοστίζουν τα κρατη Είναι κάποιο είδου βάρο για αυτού που συμμετέχουν, που απαντούν. Προσπαθούμε μόνο να καλύψουμε και αυτά τα θεματάκια. Να έχουμε εργαλεία σύγχρονα για την συλλογή των δεδομένων. Να έχουμε πηγέ διοικητικών δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα, τα αγκόρια δεδομένα, νέε τεχνικέ όπω το modeling. Transparently in the... Και επίση πω όλα αυτά γίνονται με διαφάνεια εδώ με, τη βασική, με το βασικό νομοθέτημα να ρυθμίσουμε το θέμα του κόστους μέσω του μεγέθους, μέσω της μεθόδου ε, της περιοδικότητας της διαβίβασης. Τώρα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η ευελιξία. Θέλουμε ένα πλαίσιο το οποίο να κρατήσει πολλά χρόνια. Και έχουμε τώρα ανάγκες που αλλάζουμε με ταχύ ρυθμό. Άρα χρειάζεται η ευελιξία για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις νέες απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα πρέπει να είμαστε εκεί πάρα πολύ λεπτολόγοι όσον αφορά τον κατάλογο των θεμάτων στον κανονισμό. Το αντίθετο, προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιες είδου γενικέ, γενικόλογε διατυπώσει για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Στη συνέχεια Θα έχουμε τις λεπτομερείς μεταβλητές που θα τις αφήσουμε για το τεχνικό επίπεδο. Έτσι συναρτρώνεται το πολιτικό με το τεχνικό επίπεδο. Ο νομοθέτης θα πρέπει να καθορίσει το ποια θέματα θα καλυφθούν. Οι δε στατιστικολόγοι θα συζητήσουν το πώς θα φτάσουν σε κάποιες μεταβλητές που να είναι αντιπροσωπευτικές για τα θέματα τα οποία σκοπεύουμε να μετρήσουμε. Για να υπάρχει ευελιξία λοιπόν θα έχουμε βάση του κανονισμού εφαρμοστικές και κατοξιοδότηση πράξεις. Πάντα δυνάμει της διοργανικής συμφωνίας. Τώρα, η συγκρισιμότητα. Για μας είναι από τις κορυφαίες προτεραιότητες, εκτός από το θέμα των χρονικών ε, ορίων. Χρειάζεται διαχρονική συγκρισιμότητα. Οπότε, με τις εθνικές υπηρεσίες έχουμε συζητήσει για να μην υπάρχουν διακοπές και να, και να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών. Άρα η προσέγγιση μας έχει σχέση με το αποτέλεσμα, output. Βάζουμε τους στόχους, το τι δεδομένα θέλουμε και μετά επαφείται στις χώρες για το τι input θα βάλουν για να γίνει αξιολόγηση επί τη βάση του αντικειμένου των εξολόγηση των δεδομένων. Και σας ξεκαθαρίζω ότι όταν μιλούμε για απασχόληση και ανεργία, τότε για τα δεδομένα έχουμε κάτσει και έχουμε αναλύσει εντελεχώς και καταλήξαμε στο ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ερωτηματολόγια των ερευνών. Πολλά κράτη-μέλη το είδαν έτσι. Τέτοιου είδου εναρμόνιση. Πάντω ο στόχο είναι η συγκρισιμότητα. Επίσης, στον κανονισμό θα υπάρχουν και κάποιες χρηματοδοτικές διατάξεις και έτσι οι χώρες θα μπορούσαν να αποκτήσουν τις δυνατότητες που χρειάζονται ούτως ώστε αυτή η προσέγγιση να γίνει πραγματικότητα και να έχουν επίσης κάποιες μελέτες πιλωτικές για νέα φαινόμενα και να μπορούμε κι εμείς να φτάσουμε σε κάποιες μεθολογίες στέρεες ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε για τα δεδομένα. Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να συνεργαστούμε εσείς και εμείς στενά για αυτό το θέμα. Μεγάλη μας χαρά να ακούσουμε τι σχόλια έχετε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, να συζητήσουμε, να σε εξηγήσουμε ό,τι θέλετε. Ό,τι χρειάζεται. Έτσι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να έχει καλύτερα δεδομένα τα οποία θα οδηγήσουν σε καλύτερα νομοθετήματα. Γι' αυτό και ζητάμε να μας βοηθήσετε στο έργο μας. Και ευχαριστώ. Thank you. Uh, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μέσης, κύριε Σιγητά, θα θέλετε να αρχίσετε Πρώτος με τα σχόλια. Θα ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση, η οποία ήταν σαφέστατη. Και φυσικά πιστεύω ότι οι σκιώδεις εισηγητές και όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα θα επικοινωνήσουν μαζί σας πολύ σύντομα και δεν θα περιοριστούν σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Να σας ευχαριστήσω επίσης και για τη διασφάλιση που δώσατε ότι αυτός ο εξυγχρονισμός έχει γίνει μετά από μία σειρά ε, τακτικών διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και ότι δεν είναι κάτι τελείως ε, αυθαίρετο, ούτε κάτι πρωτόγνωρο. Γι' αυτό λοιπόν δεν με εκπλήσει το αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα λιγότερο σημαντικά, μικρότερης κλίμακας, που όμως πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Και αυτό ακριβώς αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Πρέπει να ακολουθούνται φυσικά οι αρχές της διοργανικής συμφωνίας αλλά κάποιες από τις λεπτομέρειες ενδεχομένως χρειαστεί να συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό σίγουρα θα το αναφέρουν και άλλοι ευρωβουλευτές. Μετά. Κάτι σημαντικό. Ε, θα ήθελα ως εισηγητής ως αποτέλεσμα του κανονισμού αυτού να δω πολύ καλύτερη διαχείριση της ποιότητας ε, αυτών των δεδομένων που συλλέγονται και της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και επίσης να δω απόλυτη διαφάνεια στην ε, κοινοποίηση και δημοσίευση των στοιχείων αυτών. Ιδιαίτερα τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες διότι μπορεί να νομίζουμε ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αλλά πρέπει αυτή η διαφάνεια να χαρακτηρίζει όλα τα στάδια της συλλογής επεξεργασία και δημοσίευσης των δεδομένων. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε κάποια πλαίσια αναφοράς κάποια πρότυπα. Αυτό χρειάζεται ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο. Δεν είναι κάτι το οποίο, ε, με το οποίο πρέπει να επιφορτιστούν αποκλειστικά οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Οι νέες απαιτήσει, στα νέα δεδομένα θα απαιτήσουν και προσαρμογή, αλλαγή ενδεχομένως της μεθοδολογίας που ακολουθούμε. Τώρα, πόσο θα είναι αυτό το κόστος, το επιπρόσθετο κόστος. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε σύντομα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά αναπόφευκτα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την ποιότητα, για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής της άσκησης κτλ. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, παρότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν και έκανα κάποιες τοποθετήσεις που θεωρώ απόλυτα σωστές, δηλαδή για παράδειγμα για, για τη μείωση του χρόνου δημοσιοποίησης για, την, για το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται, για τους πόρους. Σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε, αλλά θα γίνει και αυτό. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τώρα λέγοντας ε, ότι αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω νομοθετήματα στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μου θα συνεργαστώ μαζί σας και προσμένω σε μια πολύ καλή συνεργασία και σε μια επιτυχημένη ε, νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πυρίνσκι και στη Λιν Κύριο Πυρίνσκι, σας ευχαριστώ. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάτι επιπλέον ουσιαστικό πω συμφωνώ με τον εισηγητή και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Μπόλεν, το ίδιο και εγώ συμφωνώ. Κυρία Λάουρενστιν, είστε και εσείς ικανοποιημένοι. Εγώ ήθελα απλώς να τονίσω ότι υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κοινωνική ε, ε, Μελέτη που δεν εντάσσεται στο σύστημα της Eurostat, αλλά ακολουθεί μια μεθοδολογία η οποία είναι απολύτως διαφανής, η οποία έχει ε, δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου και υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη βάση δεδομένων των, των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται με αυτή τη μεθοδολογία. Ελπίζω να μην το χάσουμε με αυτή τη νέα προσέγγιση της Κομισιόν. Ωραία. Μήπως θέλει το λόγο, τελευταίο λόγο, ο εκπρόσωπος της Eurostat. Ναι. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτά που ακούστηκαν και κυρίως τη γενική υποστήριξη που εκφράσετε στο προσχέδιο κανονισμού. Πιστεύω ότι η διαφάνεια και η πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα και στα μεταδεδομένα ε, είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως επίσης και το ζήτημα της ποιότητας. Όσον αφορά τη διαφάνεια. Ναι, έχουμε την πρόθεση να είναι δημοσίως διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, το ζήτημα τη συγκρισιμότητα είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό γίνεται αφενό με την εναρμόνιση των πηγών και των μεθόδων συλλογή, αφενό και αφετέρου με την ε, ε, υιοθέτηση ενό ουσιαστικού ε, πλαισίου για την ποιότητα των δεδομένων και αυτό συμπεριλαμβάνει και κάποιε εκθέσει για την ποιότητα των δεδομένων που τις μοιράζονται όλε οι αρχές, οι στατιστικέ αρχέ μεταξύ του. Η Πρόεδρος, σα ευχαριστούμε και για αυτήν την τελευταία παρέμβαση. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ε, και ήταν μάλιστα και σε, έγινε σε φιλικό κλίμα. Τη συγκρίνω με την τελευταία φορά που να συζητήσει το θέμα που είχε, ήταν αρκετά συγκρουσιακή. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Επιτροπής που ε, παρευρέθησαν και τα μέλη της Επιτροπής που παρευρέθησαν. Η συναδρίαση σήμα θα συνεχιστεί αύριο με μια σειρά ενδιαφέρον των θεμάτων. Θα ακούσουμε την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα εκπροσωπηθούν με τρεις υπουργού. Θα έχουμε επίσης την συζήτηση για την παροχή υπηρεσιών και την απόσπαση εργαζομένων. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας. Καλό απόγευμα.